πράξεις ε, σύμφωνα με την τακτική νομοθετική διαδικασία οι τίτλοι θα δημοσιευθούν στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης. Περνάμε τώρα στο